και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν από ένα χρόνο και κάτι. Το θέμα της χωριστής απαλλαγής είχε μάλιστα συζητηθεί επίσης στο πλαίσιο της υιοθέτηση του δημοσιονομικού κανονισμού, διότι είχε υποβληθεί τροπολογία από το Κοινοβούλιο για να γίνεται ξεχωριστή απαλλαγή. Κατά διάρκεια αυτής της ε, ανάγνωσης η χωριστή απαλλαγή απορρίφθηκε και προτιμήθηκε η κοινή απαλλαγή μαζί με την Κομισιόν. Από αυτή τη βάση λοιπόν εργάστηκε η Κομισιόν και διαβουλεύθηκε με μια ομάδα πυρογνωμόνων όταν εκπώνησε την έκθεση της, στην οποία συμμετείχαν και τα μέλη, μάλλον εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διανύμαμε διάφορα non-papers κατά τη διάρκεια της εξέτασης του σχεδίου ε, κατεξοδότηση πράξη και το Ελληνικό Συνέδριο εκλήθη να δώσει τις παρατηρήσεις του, να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, το οποίο και έπραξε σε ένα έγγραφο το οποίο εμείς ε, ε, υποβάλαμε και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δηλαδή και στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά και συναντήσαμε διάφορες εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ανώτερο επίπεδο και συναντηθήκαμε και με τους GTI, τους εκπροσώπους δηλαδή των ε, των, των, των συμπράξεων ε, και Πιστεύουμε πως ήμασταν απόλυτα διαφανείς στη διαδικασία με την, της κοινή απαλλαγής. Κατάλαβα τώρα πως όντως το Ευρωκοινοβούλιο ήθελε να επανεισάγει την χωριστή απαλλαγή και άρα φυσικά θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σε αυτή τη βάση. Υπάρχουν θέματα προθεσμιών και διαδικαστικά θέματα που πρέπει να αποσαφενιστούν. Αυτή τη στιγμή η περίοδος ε, ε, για υποβολή ε, αντιρρήσεων ολοκληρώνεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και αν υπάρξει αναβολή θα πάμε στην 1η Φεβρουαρίου. Αλλά επί της ουσίας είναι φυσικά μια επιλογή ανάμεσα στο άρθρο 208 που προβλέπει μέσα στην κατεξοδότηση πράξη το ίδιο το άρθρο 208 προβλέπει τη χωριστή απαλλαγή και η κατεξοδότηση πράξη είναι ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται για τις αποκεντρωμένες, ε, τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Δηλαδή υπάρχει ένα κεφάλαιο για το οποίο από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει αντίρρηση και δεν υπάρχει και συζήτηση για την κατεξοδότηση πράξη για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπάρχει επιλογή με το άρθρο 209 και τα όσα αναφέρονται στον ε, πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει να σας θυμίσω πως αυτή η επιλογή θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις πράξεις που δημιουργούν τις νέες κοινοπραξίες ή συμπράξεις και που είναι υποσυζήτηση στο Συμβούλιο και που φυσικά θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατεξοδότηση πράξη της οποίας πρόκειται εδώ και περί τη πρέπει να εργαστούμε περισσότερο είναι μια απλοποιημένη εκδοχή του δημοσιονομικού κανονισμού και κυρίως έχει στόχο να απαντήσει στις επικρίσεις ε, διοικητικού φόρτου που αντιπροσωπεύει αυτός ο κανονισμός και ο κανονισμός πλαίσιο. Αυτές οι επικρίσεις έγιναν από τους ε, ίδιους τους βιομήχανους, από τον αντιπρόεδρο της Airbus και Αυτές ε, τις δέχτηκαν οι διάφορες ε, αρχηγοί, οι διάφοροι θύνοντες των κοινοπραξιών. Εάν θέλουμε να επανεισάγουμε την κατοξιδότηση πράξη θα πρέπει να αλλάξουμε καταρχήν το δημοσιονομικό κανονισμό, το 209 και το 60, τα άρθρα 209 και 60, πρέπει να δούμε πόσο καιρό μας πάρει αυτό. Έπειτα πρέπει να μελετηθεί μια νέα κατοξιδότηση πράξη που θα υιοθετηθεί από την Κομισιόν με μια νέα περίοδο δυνατότητας έκφρασης αντίρρησης και εκεί πάλι πόσο χρόνο θα πάρει. Έχω την εντύπωση πως θα είναι δύσκολο μια τέτοια νέα ε, πράξη που θα πρέπει να αναπτυχθεί για τις ε, κοινοπραξίε ή για τις εταιρικέ σχέσεις να έχει οθετηθεί εγκαίρω όταν δηλαδή θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα νέα, οι νέες κοινοπραξίε. Μας μένει το 208, το άρθρο 208 208 ως βάση για την καταξιδότηση πράξη, για τα κοινοπραξίες που πρέπει να ξεκινήσουν τώρα. Και το άρθρο 8 ισχύει για το, από τώρα. Μας μένει το θέμα της ε, τροποποίησης των καταξιδότηση πράξεων και της εφαρμογής τους από τις κοινοπραξίες μέσα στο 2014. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα και είναι και το θέμα του να επανεξετάσουμε τι δεν πάει καλά, γιατί υπάρχουν και πολλά θετικά στοιχεία. Όλες οι κοινοπραξίες δεν είναι κατά των όσων προτείναμε, αλλά επειδή αυτά τα θέματα πρέπει να απαντηθούν σύντομα, είμαστε έτοιμοι να ε, δώσουμε όλη μας τη στήριξη για να αποσαμφωνιστούν τα θέματα αυτά συμπεριλαμβανομένων των όσων λέει ο κ. Ριβελίνη. Ευχαριστώ και συγγνώμη που με μακρηγόρησα. Ευχαριστώ δύο ομιλητέ. Τρει θέλουν να λάβουν το λόγο. Γκρέσλε, Ριβελίνη και Όντι. Ω κύριε Παραντή δεν καταλαβαίνω πολύ καλά όλα αυτά τα οποία λέτε Έγινε μια συνάντηση χθε όπου ήταν παρόντε όλοι οι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και την Επιτροπή Προπολογισμών, ο κ. Γκάιερ, ο βοηθό του κ. Γκούγεν. Και όλοι μα έχουμε κάποια δικαιώματα τα οποία δεν θέλουμε να απεμπολίσουμε. Έχουμε καταθέσει ε, τροπολογίες για τα θέματα αυτά δεν μπορούμε να χάσουμε το δικαίωμα της ε, απαλλαγής με την εξουσιοδότηση διαδικασίας. Αυτό είναι κάτι που μας απασχόλησε ήδη πριν από το καλοκαίρι. Και δεν θέλουμε λοιπόν να χάσουμε αυτό το δικαίωμα και θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια απόλυτη υποχρέωση και προς την ε, επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου και σε αυτούς που θα μας διαδεχτούν να διατηρήσουμε τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μια πληροφορία που πήρα ενδεχομένω ενδιαμέσω είναι ότι τα, οι συμπράξει αυτέ, οι κοινοπραξίε, προτιμούν να παραμείνουν στην διαδικασία αυτή του Κοινοβουλίου και όχι του, της Κομισιόν. Εμείς πάντα έχουμε απορρίψει την έννοια της ε, άμεσης απαλλαγής. Τώρα ο κύριος Σοντή Ίσως και οι συνάδελφοι τη ΣΥΤΡΑ μπορεί να δώσουν περισσότερε πληροφορίε για τα θέματα αυτά της απαλλαγή, Αλλά εμεί θέλουμε να διατηρήσουμε τη διαδικασία ω ισχύ. Μια έμεση λοιπόν για, μέσω της απαλλαγή της Κομισιόν θα ήταν μια πρόσθετη επιβάρυνση για τις συμπράξεις αυτές και αυτό νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα ε, πολύπλοκο και επιβαρυντικό για τις συμπράξεις αυτές οι οποίες θα είχαν έτσι μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο διοικητικό άχθος και δεν θέλουν επίση οι συμπράξει αυτέ να χάσουν την καλή συνεργασία που έχουν από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Εμεί επομένω καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θέλουμε να καταργήσουμε αυτέ τι εφαρμοστικέ πράξεις αλλά να αναβάλουμε την εφαρμογή τους και έχουμε προσπαθήσει με την Κομισιόν να βρούμε μια πραγματιστική λύση μας ενδιαφέρουν αυτές οι πραγματικιστικές λύσεις, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η πραγματιστική λύση μια απεμπόληση των δοκιμάτων του Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολούθησα τη συζήτηση σε σχέση με το σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού για τις ε, κοινοπραξίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα το θέμα που αφορά τη δραστηριότητα αναφοράς και τη διαδικασία απαλλαγής. Αφού συμβουλεύτηκα την Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ήθελα να προτείνω στα μέλη της Επιτροπής μας να ζητήσουμε μια παράταση του προθεσμίας για προβολή αντίρρησης ότι να εξετάσουμε καλύτερα τις πιθανές διεξόδους και το νέο πολιετές αλλά και της κατεξοδότησης πράξης. Σας ζητώ λοιπόν, μάλλον σας δίνω τους εξής λόγους για τους οποίους ε, το ζητώ αυτό. το ΕΛΚ έδειξαν αντίρρηση για την πρόταση προδιαδικασίας της τροποποίησης της διαδικασίας απαλλαγής, δηλαδή με μονομένες ε, απαλλαγές για κάθε κοινοπραξία και θεωρούν ότι αυτή η αυτή, πρόταση κανονισμού είναι ε, ζημιογόνα και καθόλου αποτελεσματική. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι η οικονομική συμβολή του ιδιωτικού τομέα και το σημαντικό ε, εφέ μόχλευση αυτή τη πρωτοβουλία απαιτεί πιο ευέλικτο δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην υπάρχει γραφειοκρατικό φόρτο και αντίθετα οι διαδικασίε να είναι ταχύτερε. Ωστόσο, πρέπει να θυμίσουμε πω το άρθρο FR 208 προβλέπει μεμονωμένη απαλλαγή αντίθετα από το άρθρο 209 που δεν το προβλέπει. Επιπλέον, το ελεκτικό συνέδριο εξέφρασε δημόσια αμφιβολίες για τη νέα διαδικασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αποτελεσματικότητα του ελέγχου, την, ορα... την ορατότητα του ελέγχου και ευθύνη. Είναι η έκθεση ε, Ρούσο. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο σε θεωρεί πως δεν ε, συμμετείχε επαρκώς στη διαδικασία διαβούλευσης για την αλλαγή του κανονισμού περί κοινοπραξιών. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε αποφασίσει με βάση το ισχύον νομικό σχέδιο, αν το συνέδριο πρέπει ή όχι να δώσει επισήμως τη γνώμη του για το θέμα. Δεν θα ήθελα εξάλλου να ξεχάσουμε πως ο Γενικός Γραμματέας του Ελεκτικού Συνεδρίου έστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης bad ε, προπολογισμού, τονίζοντας κάποιες κρίσιμες πτυχές του, του προτύπου του δημοσιονομικού κανονισμού που προτείνεται. Δεν είναι λοιπόν σαφές πώς και με βάση ποια κριτήρια οι διάφορες κοινοπραξίες θα, θα, θεωρηθούν, κοινοπραξ... θα θεωρηθούν ότι είναι συμπράξει κοινοπραξίες. Άρα λοιπόν, τίθεται σοβαρο κίνδυνο η Κομισιόν να διαλέξει με τελείως αυτόνομο τρόπο. Η νέα διαδικασία θα επηρεάσει τη μελλοντική εργασία της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και είναι άρα σημαντικό τα μέλη της Επιτροπής μας να είναι απόλυτα ενήμερα. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, η Κομισιόν θα μπορούσε να βρεθεί ενώπιον μιας, ενός πιθανού ε, ναι, είναι πιθανή, μάλλον σύγκρουση συμφερόντων. είναι ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενο, ιδιαίτερα όταν ο λογιστής τη Κομισιόν ε, ενεργεί ω λογιστή μια ή περισσότερων κοινοπραξιών. Άρθρο 22 σημείο 2. Και επίση, δεν διευκρινίζεται ποιο θα ήταν ο αντίκτυπο ε, τη διάταξη όσον αφορά την εκόρηση ενό πιο, πιο ευέλικτου δημοσιονομικού πλαισίου, ιδιαίτερα υπό το φως τη εξωτερήκευση των ελέγχων των κοινοπραξιών. Επί τη βάση λοιπόν όλων αυτών και ω εισηγητή για τον δημοσιονομικό κανονισμό θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή Κοντ μια παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων ε, και τη δημιουργία μια ομάδα ad hoc από εμπειρογνώμονες ε, της Επιτροπής Κοντ και Μπάτζ που θα αναφερθεί στα μέλη των δυο αυτών επιτροπών. Σας ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος <clears throat> Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτή την πρόταση, λέει ο κύριος Σοντή, να αναβάλουμε την εκπνοή της διαδικασίας ε, αντίρρησης. Εγώ δεν είδα όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία μας ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και προσωπικά. Θα ήθελα να αντιταχθώ στην ιδέα να ενταχθούν αυτές οι κοινοπραξίε στη γενική απαλλαγή της Κομισιόν. Είναι τόσο γενικό το θέμα αυτό που είναι ουσιαστικά δύνατο να αρνηθούμε την απαλλαγή στην Κομισιόν. Αλλά για αυτές τις κοινοπραξίες που είναι εξαιρετικές με πολύ σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτάγματα είναι πράγματι <clears throat> άξιες κάθε υποστήριξης. Και σαν μέλος Επιτροπής Βιομηχανίας τις υποστηρίζω απόλυτα. Αλλά ως μέλος τη Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και το λέω με την επιφύλαξη των διορθώσεων μπορεί να φέρει ο κύριος Ρούμπικ, ο οποίος ήταν συγκητής για τα θέματα αυτά, νομίζω ότι υπήρξαν ε, εναντί αυτών εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου, πολύ σπάνιες τέτοιες εκθέσεις, που περίχανε επιφυλάξεις. Και όταν τους ε, προσκαλέσαμε τους επικεφαλής αυτών των κοινοπραξιών, να τους εξηγήσουμε ότι τα πράγματα δεν ήταν απόλυτα εντάξει, κατάλαβαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να έχει πράγματι κάποιο έλεγχο για τα θέματα αυτά. Για τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες δίδουν σε είδος τη συμβολή τους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίδει χρήμα. Υπάρχει υποστήριξη λοιπόν για μια καλύτερη συνεργασία και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει καλύτερη παρουσίαση των συμβολών αυτών, ώστε η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να μπορέσει να ελέξει καλύτερα τις συμβολές των δύο πλευρών. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ατυχές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού ελέγχου να θέλει να αφαίρεσει από το Κοινοβούλιο αυτή την εξουσία απαλλαγής για το 208-209 δεν κατάλαβα τίποτα λέει ότι ο εκπρόσωπος Κομισιόν το 208 αφορά τον δημόσιο τομέα και το 209 τον ιδιωτικό. Μα δεν ξέρω τώρα τι, τι, τι ακριβώς γίνεται. Πότε βάζουν ένα υπόκειτο στο 208 και το 209. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο, όπως είπαν και οι δύο συναδελφοί μου, για να εξετάσουμε καλύτερα το θέμα αυτό και το Κοινοβούλιο δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο επί του προϋπολογισμού και τον πολιτικό έλεγχο σε αυτές τις δομές, ακόμα και αν είναι κούτσικο το τμήμα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού που καταλαμβάνουν. Υπήρξε η ανταλλαγή απόψεων, λοιπόν, <clears throat> μπορούμε να ψηφίσουμε για την αναβολή της προθεσμίας για την, ε, τις ποιος είναι υπέρ αυτής της ε, αναβολής, κατά, αποχές, κατά πλειοψηφία εγκρίνεται και επομένως έχει ακούσει και το μήνυμα μας η Κομισιόν. Θα, θα υπάρξει κάποιος χρόνος για περαιτέρω προβληματισμό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες προτάσεις από την Κομισιόν που να λαμβάνει υπόψη και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Εκείνη κίνηση συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού έκλεισε και ξαναγυρίσουμε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η ειδική έκθεση υπαριθμών 1 του 2013. Πρόκειται για την βιομηχανία τροφίμων με εισηγητή τον κύριο Γκέρ Μπράντι και από το ελεκτικό συνέδριο έχουμε τον κύριο Γιάν Κίνστ, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπράντι εάν προτιμάει βέβαια μπορεί να λάβει το λόγο προηγουμένως το ελεκτικό συνέδριο. Εντάξει. Παρακαλώ ξεκινήσουμε με το ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριο Κίνη, λοιπόν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω εδώ την ειδική έκθεση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή υποστήριξη στην βιομηχανία ε, τροφίμων. Να συγχαρώ τον κύριο Γκριμπράντη, ήταν πάρα πολύ καλά το έγγραφο εργασία που προετοίμασε μέρος είναι τμήμα της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν διέθεσε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2017-2013 για να ε, επενδύσει σε εταιρείε που εμπορεύονται τέτοια προϊόντα. Θεωρητικά αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να προσθέσουν αξία στα να προσθέτουν αξία στα προϊόντα προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και αυτοί οι πόροι συμπληρώνονται από εθνικές δαπάνες που ε, τελικά θρήσονται σε ύψους 9 δισεκατομμύριων ευρώ. Οι επενδύσεις ε, ε, αυτές γίνονται από καινούργιες υφιστάμενες επιχειρήσεις για μηχανήματα ή για την κατασκευή νέων υποδομών για την επεξεργασία και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Άρα το ε, ελεκτικό συνέδριο ήθελε να αξιολογήσει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αποτελεσματική στην παροχή των πόρων αυτών και κατά πόσο αυξήθηκαν η αξία των ε, γεωργικών προϊόντων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί μιλάμε για την χορήγηση πόρων σε μία από τι πιο μεγάλε και πιο ανταγωνιστικέ ε, βιομηχανίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σα πω λοιπόν ποια είναι τα βασικά στοιχεία των παρτρήσεων μα. Καταρχάς, τα κράτη-μέλη δεν απέτυξαν ότι υπάρχει ανάγκη ε, να προσμετρούνται τα προγράμματα αυτά δαπανών και αυτό σήμαινε ότι ήταν ε, επιλέξιμα πάρα πολλά τέτοια έργα στον τομέα των τροφίμων και δεν ε, εστιαστήκαμε στους πιο σημαντικούς τομείς. Το συνέδριο θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να είναι πιο συγκεκριμένα, να κάνουν μια ανάλυση κινδύνων πριν εγκρίνουν τέτοια προγράμματα, αλλά δυστυχώ έγινε μια έγκριση έτσι κι αλλιώς. Κατά δεύτερον, τα κρατημέλη δεν επέλεξαν τα έργα με, τα πιο, με το πιο υψηλό δυναμικό. Ήταν μάλλον η εξαίρεση οι κρατημέλη να ορίσουν και να εφαρμόσουν τέτοια κριτήρια επιλογής και η έκθεση παρουσιάζει παραδείγματα ατελών τέτοιων α, διαδικασιών επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιοριστήκαμε στα πιο αποτελεσματικά, πιο αποτελεσματικά έργα. Ένα άλλο σημαντικό πόρισμα του ελέγχου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν αξιολόγησαν κατά πόσο ο δικαιούχο χρειάζεται, χρειαζόταν αυτέ ε, τι δημόσια υποστήριξη, αυτό που αποκαλούμε φαινόμενο αντιπαραγωγική δαπάνη ή κατά πόσον η επένδυση βελτιώνει την κατάσταση τη εταιρεία ει βάρο ε, των ανταγωνιστών του που το ονομάζουμε φαινόμενο εκτοπισμού και δεδομένη τη ανταγωνιστικότητα του κλάδου, των αριθμών των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό ο κίνδυνο και άρα τα μέτρα αυτά ενδεχομένω ε, να βλάψουν τελικά την βιομηχανία. Όλες αυτές λοιπόν, όλα αυτά τα ελαττώματα, όλε αυτές οι ατέλειε ε, εξηγήθηκαν στην ανάλυση του συνεδρίου και όπως σας εξήγησα Το θέμα ήταν να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία και να μην υπάρξει αυτό το φαινόμενο αντιπαραγωγική ε, δαπάνη, να μην υπάρξει το φαινόμενο του εκτοπισμού. Ωστόσο, σε δύο μόνο από τα 24 έργα θεωρούμε ότι πληρούνται τα κριτήρια αυτά. Σε 10 εξ αυτών πληρούνται κάποια από αυτά τα κριτήρια. Θα έπρεπε να τονίσουμε ωστόσο ότι η επιτυχία των έργων αυτών δεν ε, έχει να κάνει τόσο πολύ με τα συστήματα επιλογής που εφαρμόστηκαν από τα κρατημέλη, γιατί τα, πολλές φορές τα ίδια κρατημέλη εμ, έδωσαν τέτοιους πόρους σε άλλα 12 έργα, τα οποία θεωρούμε ότι δεν ήταν αποδοτικά. Τέλος, το συνέδριο θεωρεί ότι τα κρατημέλη δεν ε, επιτήρησαν, δεν παρακολούθησαν επαρκώς τα αποτελέσματα του project. Θα ήθελα να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι το συνέδριο πριν από κάποιες εβδομάδες ενέκρινε ένα ειδικό έλεγχο σε ό,τι αφορά ε, τέτοιες αξιολογήσεις, σε ό,τι αφορά προγράμματα ανάπτυξης της υπέτρου. Θα χαρώ να σας παρουσιάσω τα απορίσματα αυτά. Το συνέδριο λοιπόν επίσης παραχύει τις συστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κρυμπράντη που είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ τον κύριο Κίνς για τη σαφήνεια των εξηγήσεων που μας έδωσε. Μόνο οι δυο μας ουσιαστικά τώρα έχουμε μείνει σε αυτή την αίθουσα. Μήπως μπορώ να, ψηφίσω, να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση σε λίγο. Μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Μπορεί, να πάρω διαφορετική θέση από εσά, οπότε θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. το σκεφτώ, λέει ο κύριο Κερμπράντη σε πιο σοβαρό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε ένας στην Ευρώπη, ο οποίος αφού διαβάσει την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, που θα έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουμε αμέσω τα μέτρα 1, 2 και 3. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε την επόμενη εβδομάδα. Είδα πολλές ειδικέ εκθέσεις από το ηλεκτρικό συνέδριο. Πολλές από αυτές είχαν ανησυχητικό χαρακτήρα. Αλλά αν δω τώρα τα συμπεράσματα και τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου για το μέτρο αυτό το 1-2-3, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουμε στην Ευρώπη με 5,6 δισεκατομμύρια χρημάτων των φορολογουμένων. Για να τα πω απλά, δεν υπάρχουν κάποιοι στόχοι επί τη βάση των οποίων μπορούμε να καταμετρήσουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών μας. Απλώς πρόκειται για μια γενικευμένη αγροτική ανάπτυξη για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Και με τέτοιο γενικό στόχο εμείς δίνουμε 5,6 δισεκατομμύρια σε εταιρείε και μάλλον μεγάλες εταιρείε οι οποίες θα μπορούσαν οι ίδιες να χρηματοδοτήσουν τις ενέργειές τους το βρίσκω λίγο απίστευτο. Η νομοθεσία δεν αναφέρει καθόλου ποια είναι η προστοκόμενη προσθέμενη αξία. Ούτε καν ζητάμε λοιπόν για προσθέμενη αξία, απλώς θέλουμε να δαπανώνται τα χρήματα. Και παραθέτω αυτό που αναφέρεται εδώ. Ο στόχος, ο μόνος στόχος ο οποίος επιζητείται είναι να υπάρξει κάποιο όφελος προς τις συγκεκριμένες εταιρείες εμπορίας καρπών. Μα όταν δίνετε λεφτά πάντα είναι ευχαριστημένες οι εταιρείε αυτές. Δεν ξέρω λοιπόν τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο να δίνουμε τόσα λεφτά. Το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει ε, εντοπίσει συγκεκριμένες ανάγκες για παρέμβαση στον τομέα μεταποίησης τροφίμων, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να δοθούν τα χρήματα αυτά. Δεν υπάρχει ορθολογικός αποχρόν λόγος για τα μέτρα αυτά. Δεν έχουμε κανένα λόγο για να πάρουμε αυτά τα μέτρα, δεν έχουμε κανένα στόχο επί τη βάση του οποίου να μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο επιτυγχάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε και παρόλα αυτά δίνουμε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και δεν τελειώνει εδώ το θέμα γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Μέσα στην τρέξα δημοσιονομική περίοδο είδαμε τα προβλήματα αυτά. Στην προηγούμενη φορά ήταν κάπως καλύτερα, αλλά έχουν γίνει χειρότερα. Και τώρα εν ώψη των προτάσεων για την επόμενη ε, περίοδο χρηματοδότησης δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως κοινοβούλιο ενώπιον μιας τέτοιας τόσο συντριπτικής έκθεσης από το ελεγκτικό συνέδριο. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτές τις επικρίσεις μέσα στον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου. Είδαμε τα ίδια με το αγροτοπεριβαλλοντικό σχέδιο, όπου και πάλι υπήρξε μια συντριπτική ανάλυση εναντίον του από το ελεκτικό συνέδριο. Προσπάθησα να θέσω στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 10% αυτών των ποσών στο αποθεματικό. Απέτυχα γιατί οι περισσότεροι δεν θέλαν να μπουν στο αποθεματικό. Και το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω είναι να κάνω μια σύνδεση μεταξύ στόχων και κονδυλίων που θα πρέπει να γίνεται για οποιαδήποτε γραμμή του προπολογισμού. Αλλά φαίνεται ότι, και αυτό είναι σαφές και από την ετήσια έκθεση του 2010, 12 παρουσιάστηκε πριν από δύο μέρες εδώ, η καταβολή των κονδυλίων είναι πιο σημαντική από το να εξετάσουμε τι σκοπό εξυπηρετούν τα κονδύλια αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα βέβαια. Το νομοθετικό πακέτο για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο είναι κοντά στο, στην οριστική του έγκριση. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να αφήσουμε να περνάει ένα τέτοιο μέτρο. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ, και αυτή είναι και η πρώτη σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου, και εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Το ερώτημα μου προς η Κομισιόν είναι, η Κομισιόν είναι έτοιμη να εγκρίνει μόνο αυτά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από τα κράτη-μέλη που έχουν τεκμηριωμένες και ουσιαστικές στρατηγικές με ορθολογική βάση για να δείξουν πώς αυτή η χρηματοδότηση θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Φοβάμαι ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο. Εάν δεν το κάνει η Κομισιόν, εγώ δεν έχω καμιά άλλη επιλογή, αλλά να προσπαθήσω να θέσω όχι το 10% αλλά το σύνολο της γραμμής αυτής του προϋπολογισμού στο αποθεματικό του χρόνου. Κλείνω εδώ και δεν ξέρω αν μπορούμε μαζί με τους συντονιστές, αυτό θέλω να σας ρωτήσω εσάς κύριε Πρόεδρε, αν μπορούμε μαζί με τους συντονιστές να βρούμε τρόπους για να καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα καταρχάς να υποδείξω ότι ο αριθμός ε, των <laughs> μελών έχει αυξηθεί κατά 50% και ήρθε και ο συνάδελφος Γκάι. Μάλιστα, ναι. Μπορούμε να πάμε να πιούμε καφέ και να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις μας μεταξύ μας. Έχουμε value for money σε αυτή την περίπτωση. Ένα πράγμα που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Υποστηρίζω όλα όσα μας είπε ο συνάδελφος και ευχαριστώ το λεκτικό συνέδριο. Είμαι αρμόδιος ε, για τα σύνορα τα Ολλανδικά, τα Γερμανίες με την Ελλανδία και διαπίστωσα τις με μεγάλη έκπληξη ότι ο μεγαλύτερος αποδοχέας γεωργικών πόρων είναι η εταιρεία Κατσίς. Παράγει πόσιμο νερό και θα τα γνωρίσετε. Το τελευταίο πρόβλημα που έχει αυτή η εταιρεία, εν περιπτώσει, είναι ρευστότητα. Καλό είναι βέβαια αυτό για την εταιρεία, αλλά γιατί πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατάσταση τη εταιρεία αυτή, ε, δίδοντα ευρωπαϊκού πόρου, εγώ τι να σα πω, δεν το καταλαβαίνω. Και ε, πολύ σωστά διαπιστώνει το εκτικό συνέδριο ότι τα κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις δεν νοιάζονται για το κατά πόσον οι εταιρείε που τελικά λαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς πόρους τους χρειάζονται όντω για την καινοτομία. Το θέμα είναι να κυλάει το χρήμα. Αυτό ισχύει τουλάχιστον στη Γερμανία. Και δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο παράδειγμα αυτό που αναφέρω. Και γι' αυτό λοιπόν ε, δεν ε, συμφωνώ με τον κύριο Κλίντς που λέει ότι υποχρεούνται να κάνουν το οτιδήποτε. Αυτά προκαλούν την κατάσταση, είναι στον πυρήνα του προβλήματος. Και δεν ξέρω πώς ε, μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Και θα πρέπει, δεν χρειάζεται να σας αναφέρω εδώ, πόσο σημαντικό είναι το λόμπι των γεωργικών προϊόντων εδώ στο Κοινοβούλιο. Και δυστυχώς αυτό αφορά και την δική μου την ομάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια. Καταρχάς λοιπόν, θα έλεγα ότι τα πορίσματα αυτά θα πρέπει να τα θίξουμε εδώ στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την χορήγηση της απαλλαγής. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Πολύ πιο σημαντικό ίσως και από πολλά άλλα θέματα τα οποία το τμήμα του τριδουργικού. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να περάσει στην Ολομέλεια και θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους συντονιστές κατά πόσον θέλουμε να είναι η έκθεση αυτή ή κατά πόσον θα δημορφωθεί ως ερώτημα. Στην Ολομέλεια πάντως να πάει. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κατα ποσον θα δημιουργηθει ως ερωτημα στην ολομελεια παντως να παει θα ειναι παρα πολυ ενδιαφερουσα η συζητηση Σας... Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάιερ υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν κατά πόσο θέλει να λάβει θέση σε σχέση με αυτά. Κύριε Σούσα, ούβε, έχετε το λόγο εφόσον θέλετε να αναφερθείτε στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, εκπροσώπους της ε, Επιτροπής σας και του Ελεκτικού Συνεδρίου Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ορισμένα στοιχεία που νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το μέσο, αυτό. Ο εισηγητής μου έθεσε ένα σαφές ερώτημα. Κατά πόσον δηλαδή υπάρχει μία ε, εξέλιξη η οποία οδηγεί σε πιο στοχευμένο μέτρο. Όλη η λογική μας στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα είναι να εστιάσουμε καλύτερα το μέτρο αυτό και να εστιάσουμε καλύτερα στις έξι προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές που έχουν ε, να κάνουν με τα μέτρα για την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας. Αναφέρουμε λοιπόν στις προτεραιότητες 2 και 3 του μελλοντικού κανονισμού και στα μέτρα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18 του προσεχούς κανονισμού και επίσης σε κάποιο βαθμό στο άρθρο 20 του επικείμενου κανονισμού για την καλύτερη εστίαση στην ανταγωνιστικότητα και και την υποστήριξη των δικαιούχων. Βρισκόμαστε πάντα σε μια διαδικασία διαμερισμένης διαχείρισης. Τα κάτι μέλη θα φέρουν μια στρατηγική θα έχουν τις ανάγκες οι οποίες θα έχουν εντοπιστεί σε αυτή, στα πλαίσια της στρατηγικής και θα παρουσιαστούν προγράμματα τα οποία ε, καθορίζουν τις ανάγκες της κάθε περιοχής και τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να εστιάσουν περισσότερο στις ανάγκες αυτής της περιοχής σε ποσοτικό επίπεδο. Και όλα αυτά θα μετρώνται σταδιακά μέσω ενός πλαισίου αξιολόγησης που βασίζεται σε δείκτες αποτελεσμάτων που θα είναι και αντικτύπου που θα πρέπει να μετρούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Άρα λοιπόν, ε, Αυτά λοιπόν όλα με βάση συγκεκριμένους στόχους ε, για τα διάφορα μέτρα. Επιτρέψατε μου όμως, ε, αφού ξεκίνησα με μια άμεση απάντηση προς το ερώτημα που υποβάλλατε, επιτρέψατε μου ωστόσο να σας δώσω και το συγκεκριμένο μέτρο ε, στο πλαίσιό του. Διότι θα ξεκινήσω λέγοντας πως η ε, έννοια, μάλλον η σύλληψη αυτού του μέτρου είναι προστεθέμενη αξία για τα γεωργικά προϊόντα. Αλλά η αντίληψη του 1698, η νομοθετική, είναι πολύ ευρύτερη, γιατί εκεί περιλαμβάνεται η, προσ... η, η, η πραγματική αξία μέσω της λήψης υπόψη των βελτιώσεων στο επίπεδο της διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος, επίσης των πτυχών που έχουν σχέση με την διατροφική ασφάλεια, την ε, διατροφική υγεία, αλλά και την ευημερία των ζώων. Μπορεί να συμφωνεί κανείς, αλλά μπορεί και όχι. Ο νομοθέτης έτσι το έχει ορίσει, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής αυτού ε, του μέτρου. Είναι μια διάσταση αυτή την οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν κρίνουμε το μέτρο. Η προσδεθέμενη αξία λοιπόν θα πρέπει να μετράτε με διάφορα μέσα στήριξης για τα διαφορετικά είδη χρηματοδότησης που θα μετρούν την αποτελεσματικότητα, την προώθηση των μεταποιημένων προϊόντων στο πεδίο όχι μόνο της διατροφικής αλυσίδας αλλά και της ανανεώσιμης ενέργειας καθώς επίσης και μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών που ε, ε, ε, διανοίγουν νέες ευκαιρίες για την αγορά, αλλά και σε σχέση με την διάσταση της ποιότητας. Και υπογραμμίζω όλες αυτές τις πτυχές ώστε να τονίσω πως το πεδίο εφαρμογή του μέτρου είναι ευρύ. Έπειτα, κύριε Πρόεδρε, ο νομοθέτης ε, έχει δει να εξελίσσεται αυτό το μέτρο διαχρονικά αφήνοντας το κράτος μέλος την δυνατότητα να ανοίξει το πεδίο, διευρύνει το πεδίο χρήσης του μέτρου. Είναι σαφές κύριε Πρόεδρε ότι σε θέματα επιλογής Στη νέα περίοδο, στο άρθρο 49 του νέου κανονισμού, η Κομισιόν υποβάλλει νέα πρόταση, μέσω της οποίας εισάγονται κριτήρια επιλογής, που τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά. Ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε κύριε Πρόεδρε πως ε, υπάρχουν διάφορες ε, πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή των ε, προγραμμάτων. Όταν η Κομισιόν εγκρίνει τα προγράμματα και όταν προβαίνει σε αξιολόγηση του προγράμματος και των μέτρων, οφείλει να αναλύσει την σύσταση τους και την στρατηγική, όπως ήδη σας ανέφερα, αλλά πρέπει να δει επίσης πως κατά πόσο μάλλον το μέτρο αυτό έχει κατάλληλο στόχο και αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ξεκάθαρους στόχους που ανταποκρίνονται σε διαρθωτικές ανάγκες και σε εδαφικές ανάγκες. Και, αυτός, και αυτή η στοχοθέτηση στη συγκεκριμένη περίοδο έχει επιτευχθεί είτε μέσω των κριτηρίων επιλογής είτε μέσω των όρων επιλεξιμότητας είτε μέσω της διαφοροποίησης των ενισχύσεων σε διάφορα επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη το είδος του αποδέκτη, το είδος της επένδυσης και το επίπεδο Στήριξη και κριτική ενίσχυση. Όλε αυτέ αυτές οι επιτυχίες λοιπόν αποτελούν παράγοντες που στόχο έχουν τη στοχοθέτηση του μέτρου στην υπηρεσία ενός, μιας υπηρεσίας και αρχικής στρατηγικής. σας ζητώ λοιπόν όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη και να μην ε, εξετάσετε μόνο αυτό το μέτρο ότι εξυπηρετεί άνευ κριτηρίων αποδέκτες ανεφορίων. Είναι ένα σύνολο δηλαδή που στόχο έχει τον παραλήπτη μέσα στο σεβασμό του πνεύματος του νομοθέτη του 2015 όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός 1698. Τώρα παραμένουμε σε αυτή την ε, κατάσταση ή προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη στόχευση. Σας παρακαλώ λοιπόν να θεωρήσετε θετική την απάντησή μου. Ναι, προχωρούμε προς καλύτερη στοχοθέτηση. Πώς? Μέσω μιας στρατηγικής ενισχυμένης που ορίζει το σχέδιο του προγράμματος είναι πιο συγκεκριμένη όσον αφορά τα θέματα επιλογής και, και επιλεξιμότητας Επίσης υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην, στο είδος στήριξης και στην ένταση της στήριξης που δίνεται στο άρθρο 18 και κυρίως ενισχύοντας την ανίσχυση απόδειξης. Δηλαδή, με ποιον τρόπο το μέτρο processing και marketing συμβάλλει στους στόχους της στρατηγικής και ποια μέτρα συγκεκριμένα ε, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται μια προσπάθεια στόχο έχει να ανταποκριθεί στις ανησυχίες αλλά και στις αδυναμίες που εντοπίζονται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης, ε, θα υπάρξει συνοδευτική προσπάθεια ανάλογα με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει και τις απαιτήσεις που έχουν εισαχθεί στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αυτό το συνοδευτικό σύστημα παρακολούθησης δηλαδή και ελέγχου και αξιολόγησης έχει στόχο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τα, για να μετρήσουμε καλύτερα την αποτελεσματικότητα του μέτρου που εξυπηρετεί τις δύο προτεραιότητες, την αντιγνωστικότητα της ε, αγροδιατροφικής αλυσίδας. Με δύο λόγια λοιπόν, αυτά είχα να σας πω ως στοιχεία που βελτιώνουν το μέτρο, διότι ο νομοθέτης σε μια διαδικασία συναπόφασης ε, βρήκε τη συνένεση γύρω από αυτή την νομοθετική πρόταση που φυσικά υπόκειται στην έγκριση του Κοινοβουλίου αλλά που τονίζει τη βελτίωση της πολιτικής της ανάπτυξης υπαίθρου ώστε να επιτευχθεί η αντικειμενικότητα ε, και έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία της διατροφικής αλυσίδας όταν μιλάμε πια για τη φάση της βιομηχανίας μεταποίησης. Επιστήνονται την προσοχή σας στο γεγονό ότι στα άρθρα 18 και 20 της νέας πρότασης ο σύνομοθέτης έχει ε, ορίσει ένα πλαίσιο όπου η διάσταση του ε, αποδέκτη ε, λαμβάνεται υπόψη ώστε να εστιαστεί στις ανάγκες της κατάλληλης διάστασης. Για το θέμα του The Θέλω να σας πενθυμίσω στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη διευκρινίσουμε ότι για τις αγροτικές ε, δαπάνες μία δαπάνη που γίνεται μετά από την υποβολή των αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές θα θεωρηθεί ότι είναι ε, επιλέξιμη και τα λέω στα αγγλικά για να παραμείνω μέσα στα πλαίσια του κτηρίου του, του κειμένου καλύτερα το οποίο έχει εγκριθεί με γενική συνένεση τα λέω αυτά για να κατανοήσετε ότι θεωρούμε ότι υπάρχει με τον τρόπο αυτό ένα στοιχείο παρότρινσης από το οποίο αποτρέπει του κίνδυνος αυτός. Και έχουμε λοιπόν μια στρατηγική η οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό και είναι προς το συμφέρον μας να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έχουν υπογραμμιστεί και από το Ελληνικό Συνέδριο για να αποτρέψουμε τα στοιχεία του εκτοπισμού και έτσι η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει στην έκθεση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή και το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Σας ευχαριστώ για την ε, <clears throat> παρέμβασή σας. Ελπίζω Ελπίζω μην εφαρμόζεται ένας κανόνας από τις προηγούμενες δραστηριότητές μου που είχα τότε διαπιστώσει ότι όσο πιο μακρά είναι μια παρέμβαση, τόσο λιγότερα πράγματα λέει και τόσο λιγότερες αλλαγές αντανακλά, λιγότερη θέληση αλλαγής. Ελπίζω λοιπόν θα λάβετε υπόψη την θέση του ελεκτικού συνεδρίου στα σοβαρά και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή αν θέλει να προσθέσει κάτι σε όλα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εγώ το σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την έκταση της παρέμβασης και την προθυμία να αλλάξει πραγματικά κάτι. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, σε μένα με ανησυχεί πιο πολύ η κατάσταση. Τώρα μετά την απάντηση, γιατί θεωρώ, θεωρούσα ότι η Επιτροπή ήταν εταίρος μας, εταίρος του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της ε, σωστής δαπάνης των ευρωπαϊκών πόρων και στην αναζήτηση ε, τρόπων αύξησης της υποστήριξης του κοινού για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι αυτός τρόπος να προχωρήσουμε. Μία σύγκριση. Έχουμε το χρηματοοικονομικό μέσο για την ε, φύση. 3,8 δις. το Nature. Έχουμε διάφορες εκθέσεις, τριμερή διάλογο, μια τεράστιο καυγά που έγινε με το Συμβούλιο για όλα τα στοιχεία της νομοθεσίας. Και μιλάμε για το 60% του μέσου αυτού. Γιατί εδώ μιλάμε για 5,6 δισεκατομμύρια. Και εδώ δεν φαίνεται καν να αναρωτιόμαστε γιατί τα ξοδεύουμε μετά τα χρήματα αυτά. Ναι, εντάξει, να μιλήσουμε για στοχευμένη προσέγγιση, για ποσοτικοποιημένα μέσα, για το άρθρο 18 του επόμενου κανονισμού, για τη συμπερίληψη μέτρων για ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, αλλά και πάλι το Συμβούλιο αμφισβητεί την ύπαρξη του μέσου. Δεν υπάρχει φαίνεται καν κάποιος λόγος για να υπάρχει αυτός, αυτό το μέσο και για να ταπανώνται τα 5,6 δισεκατομμύρια τα επόμενα 7 χρόνια στην ε, βιομηχανία τροφίμων. Όπως είπα λοιπόν, πλέον δεν ξέρω τι να σας πω, ανησυχώ πιο πολύ από ό,τι ανησυχούσα πριν από την συνάντηση αυτή, πριν από τη συνεδρίαση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει περίπτωση να κάτσει να αναρωτηθεί εκ νέου γιατί το κάνουμε αυτό γιατί πανώ με τα κονδύλια αυτά. Ή τουλάχιστον να ζητήσει από τα κράτη-μέλη στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου να μην εντοπίσουν μόνο τους λόγους για τους οποίους ε, χορηγούν τα κονδύλια, αλλά και το τι ελπίζουν να πετύχουν με τα κονδύλια αυτά. Φυσικά, η κοινή διαχείριση και άλλες τέτοιες εκφράσεις πάντα μου αρέσουν, αλλά είμαστε ρεαλιστές. Τα κράτη-μέλη δεν νοιάζονται για το πού πάνε τα λεφτά. Αυτό που τα απασχολεί είναι να πάρουν από το κουμπαρά των Βρυξελών όσο πιο πολλά χρήματα γίνεται για τη χώρα τους. Αυτό τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ αυστηρές ε, διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πού θα πρέπει να πηγαίνουν τα κονδύλια αυτά. Όχι, σαφείς στόχους θα πρέπει να έχουμε. Και σαφείς τρόπους να τα πετύχουμε αυτά. Ιδάλλως να ζητάμε συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Γιατί δεν πετύχαμε τους στόχους μας. Και ιδάλλως να κάτσουμε να σκεφτούμε κατά πόσο θέλουμε να συνεχίσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό περιμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως να μην κατάλαβα όλα όσα είπατε. Διάφορα άρθρα στα οποία αναφερθήκατε. Ειλικρινά δεν τα ξέρω απ' έξω. Ίσως να κρύβεται κάπου αλλού λοιπόν η ουσία του θέματος. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν μου διαφεύγει κάτι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι καλά θα κάναμε να ακολουθήσουμε την πρόταση του Γιάνν Γκάιερ να περάσει στην Ολομέλεια το θέμα, είτε με έκθεση είτε με ερώτημα προφορικό. Αλλά σας παρακαλώ πρόεδρε, συζητήστε το με τους συντονιστές να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Ε, ναι, Πολύ ευχαρίστω θα ακολουθήσω την πρόταση των συντονιστών. Θα του θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, την κοινή επιχείρηση Excel. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κάιερ. Αγαπητέ Μιχαέλ, αγαπητέ Γιάννη, τώρα είμαστε σε οικογενειακή φάση. Δεν μπορώ να πω τώρα Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είμαστε τόσο λίγοι. Πρόκειται για μία νέα σύμπραξη η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση των προηγουμένων ενεργειών μια πρωτοβουλία η οποία θα βοηθούσε την νανοτεχνολογία, την Άρτεμι και μια άλλη η οποία αφορά τα εν, ε, ενσωματωμένα συστήματα ο στόχος είναι να υπάρξει μια νέα κοινή ε, πρωτοβουλία που λέγεται Excel, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το πρόγραμμα πληροφορικής. Εμείς πρέπει να δώσουμε μια γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά προς την Επιτροπή Ήτρα, η οποία είναι η αρμόδια επί της ύλης. Το έχω πράξει αυτό με την ε, βοήθεια της γραμματείας. και έχω προσπαθήσει να παρουσιάσω τη δική μας άποψη σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την ε, απλοποίηση των ε, ε, ιδιωτικών επενδύσεων σε συνεργασία με δημόσιες επενδύσεις και φυσικά δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε πολιτικό επίπεδο για μια τέτοια πρωτοβουλία από τον εκτελεστικό διευθυντή της Excel έγινε σαφές ότι εμείς θα πρέπει να συμμετέχουμε πλήρως σε αυτή τη διαδικασία, ότι πρέπει να αποτραπούν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι ο ελεγκτής της ε, Κομισιόν θα συμμετέχει στην έκθεση υπεπραγμένων της Excel ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ότι θα υπάρξει και δήλωση των ε, οικονομικών συμφερόντων του Διοικητικού Συμβουλίου της Excel ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να αποτραπούν ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Μετά από αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης, δηλαδή για τις νομικές διατάξεις που βρίσκονται στον κανονισμό για τις ε, συμπράξεις, να συμμορφωθούμε και έχουμε ήδη ακούσει τις προτάσεις στον τομέα αυτό από πολιτική άποψη. Δεν είναι ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα και γι' αυτό δεν περιμένω ότι θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, αλλά είμαι φυσικά ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση των συναδελφών. Ευχαριστώ πολύ, λέγει ο πρόεδρος. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο, Όχι, ο Γιάν. <clears throat> Ήταν ενδιαφέρον πάντως το ζήτημα αυτό και ευχαριστώ τον κύριο Γκά για την ε, παρέμβασή του. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, κύριο Γκλοκ Γκλουκ, όπως λέγεται, και να στήσω και την άποψη της Κομισιόν. Ε, thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά ε, την ε, σύμπραξη αυτή και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Artemis. Ε, αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων συνεργειών στα πλαίσια του Excel. Υποστηρίζουμε την πρώτη τροπολογία που ζητά απλοποιημένο μοντέλο λειτουργίας και σχετικές απλοποιημένες διαδικασίε. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάζεται κατεπηγοντός σε αυτόν τον τομέα του Excel σε ό,τι αφορά τα ευφύ e συστήματα, τα ενσωματωμένα μικροελεκτρονικά συστήματα. Για τις άλλες τροπολογίες, να σας πω ότι προβλέπεται να υπάρξει ικανότητα εσωτερικού ελέγχου αυτό ενδεχομένω να επηρεάσει τις ε, τροπολογίες και σε ό,τι αφορά τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή. Αυτό το επεξεργάζεται και το καταστατικό της ε, κοινοπραξίας Excel. Άρα, ναι, καλωσορίζουμε αυτή την έκκληση για απλοποιημένους όρου λειτουργίας, προκειμένου και ο κλάδος να μπορέσει να ανταποκριθεί πολύ ταχαίως σε έναν ανταγωνισμό μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο με τις άλλες περιφέρειες. Είναι πραγματικά αμήλικτος ο ανταγωνισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την παρέμβασή σας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε στην παρούσα φάση και ως εκ τούτου νομίζω ότι ολοκληρώσαμε σε περίπτωση τουλάχιστον που ο εισηγητής δεν θέλει να πάρει το λόγο. Θες να πεις τίποτα, ναι, όχι, όχι, να το κλείσουμε. Μάλιστα, ναι, κάπως και εγώ επιτάχυμα τις διαδικασίες προκειμένου να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ελεκτικού Συνεδρίου, της Γραμματείας, τους Διερμηνείς και όλους όσοι μας βοηθήσαν σήμερα και έτσι λοιπόν κλείνει τη σημερινή συνεδρίαση στις 7 Νοεμβρίου. Καλό βράδυ και καλή επιστροφή σε όσους ε, έχουν ταξίδι μπροστά τους. Ευχαριστώ πολύ.